Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, dear colleagues. Welcome to... αγαπητοί συνάδελφοι. Καλώ ήρθατε στην ε, συνεδρίαση τη Επιτροπή μα. Ε, είναι 9 και 7 λεπτά ολόκληρα, οπότε α ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Περνάμε στο σημείο 13 της ημερησίας διάταξης ε, και πάλι, μας, πάλι με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε τον κύριο Ιωάννης Χάν, Επίτροπο Πολιτικής ε, γειτονίας και διεύρυνσης στην Επιτροπή του, την Επιτροπή των Εξωτερικών. Ε, θα θέλαμε να συζητήσουμε ακόμη μια φορά και ελπίζουμε τελευταία φορά με τον κύριο Χάν ε, ζητήματα διεύρυνσης και γειτονίας. Λοιπόν, θα αντιστρέψουμε την συνήθι σειρά και θα ξεκινήσω ευχαριστώντας σας αγαπητέ Γιωχάνες εξ ονόματος της Επιτροπής μας για την συνεργασία που είχαμε και για τις άοκνες προσπάθειές σας να καταστήσετε επιτυχή την θητεία που μόλις πέρασε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να έχουμε και με την διάδοχό σας ε, εξίσου καλή συνεργασία. Και βεβαίως ε, έχουμε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή, όπως και άλλοι συνάδελφοι στην αίθουσα. Έτσι και εγώ ήμουν πολύ όμως ε, και έλεγα πως ε, το ότι δεν ελήφθη απόφαση για Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία ήταν μια κακή μέρα για την Ευρώπη. Δεν προωθήσαμε τη συμφιλίωση στην Ευρώπη. Απογοητεύσαμε τους συμμάχους μας και επιδείξαμε έλλειψη στρατηγικού οράματος. Και αυτό λόγω μιας ε, ελάχιστης μειοψηφίας ε, κρατών μελών. Νομίζω ότι πρέπει να αποστείλουμε σαφή μηνύματα, ειδικά στα Σκόπια, ότι θα τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας και δεν θα προδώσουμε τους φίλους και συμμάχους. Να πω ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριος Σασόλη, ήδη έχει πάει στην Βόρεια Μακεδονία για την ε, πρώτη του επίσκεψη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως θα ακολουθήσει και στις 2 και 3 Δεκεμβρίου η επίσκεψή του στην Αλβανία. Τέλος πάντων, ό,τι έγινε έγινε. Ας δούμε τώρα τι μπορούμε να κάνουμε για να προετοιμαστούμε για την ε, διεύρυνση, για να μην μείνουν όλα αυτά κούφια λόγια. Οπότε ας δούμε και τις προκλήσεις στην ευρύτερη γειτονιά μας. Αγαπητέ Γιωχάνες, θέλουμε να ακούσουμε τις απόψεις σας, όχι μόνο για την κατάσταση στα Βαλκάνια, αλλά και για τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας, ειδικά Γεωργία, Μολδαβία και Ουκρανία. Επίσης, να ακούσουμε και τα σχέδιά μας για αναθεώρηση αυτής της πολιτικής μετά από 10 χρόνια. Τέλος, να τονίσω την σημασία της επαρκούς χρηματοδότησης και σεβασμού των προνομίων του Κοινοβουλίου όσον αφορά την χρηματοδότηση της εξωτερικής πολιτικής δράσης και τη προενταξιακή ε, βοήθειας. Οπότε καλώ ήρθατε και πάλι κύριε Επίτροπε στην Επιτροπή μας ε, και η συζήτηση μαζί σας ε, θα κρατήσει μέχρι τι 10 και μετά θα συνεχιστεί ως στρατηγικός διάλογος. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Νταβίντο. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία την τελευταία πενταετία με πολλούς από εσάς ε, και με την ε, ενεργό σε συμμετοχή προσπαθούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση στη γειτονία μας, ε, την πιο κοντινή και την πιο μακρινή. Εισαγωγικά θα ήθελα να επικεντρωθώ στα Δυτικά Βαλκάνια, διότι αυτή τη στιγμή εκεί έχουμε την ε, πιο σημαντική επικαιρότητα. Ίσως, όπως είπατε, να είναι η τελευταία μου ε, ομιλία εδώ στην Επιτροπή σας. Ε, όταν ανέλαβα καθήκοντα το 2014, η κατάσταση ήταν δύσκολη. Είχαμε ακούσει την φημισμένη δήλωση του Πρόεδρου Γιούνκερ που πολλοί δεν κατάλαβαν σωστά ότι δεν έπρεπε να γίνει άλλη διεύρυνση. Όποιος γνωρίζει τα θέματα όμως ε, κατάλαβε τι εννοούσε, αλλά πολύ τότε το παρανόησαν. Από την ε, αρχή προσπαθούσαμε να πούμε πολύ σαφώς, πολύ καθαρά ότι υπάρχει μια σαφής ευρωπαϊκή προοπτική για όλες τις ε, χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που ακόμα δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας συνοψίσω για λίγο τι σημαίνει αυτή η σαφής προοπτική, τι σήμαινε τα τελευταία πέντε χρόνια και τι δυνατότητες έδωσε. Πρώτα απ' όλα έδωσε τη δυνατότητα όπως ε, αναφέρεται στη στρατηγική μας του 2008 για τα Δυτικά Βαλκάνια, μια νέα χώρα μέλος μπορεί να γίνει μέλος ε, όταν όλες οι διμερείς διαφορές ε, έχουν επιληθεί πριν γίνει μέλος. Και αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να γίνουν πολλέ συζητήσει, ώστε να επιλύσει για παράδειγμα η Βόρεια Μακεδονία τη διένεξη με την Ελλάδα που είχε διαρκήσει δεκαετίες να έχει μια συμφωνία με την Βουλγαρία το Κωσυφοπέδιο και το Μαυροβούνιο να επιλύσουν το εκρεμή ζητήματα των συνόρων. Όλα αυτά έγιναν δυνατά ε, λόγω της ευρωπαϊκής, σαφούς ευρωπαϊκής προοπτικής. Από την αρχή, βάσει της διαδικασίας του Βερολίνου, ε, από το 2014, που ξεκίνησε το 2014 επικεντρωθήκαμε έντονα στην περιφερειακή ανάπτυξη με τα αντίστοιχα προγράμματα. Κατά μέσο όρο ετησίως ε, δώσαμε, επενδύσαμε σχεδόν ένα δισεκατομμύριο ευρώ στα Δυτικά Βαλκάνια και μιλάω συνειδητά επενδύσεις, όχι απλά επιχορηγήσεις. Από την άλλη πλευρά ε, το πρόγραμμα του Βερολίνου προωθεί την περιφερειακή ανάπτυξη και την εφαρμογή της στον τομέα της συνδεσιμότητας, υποδομές, ε, μεταφορές, ε, αλλά και στον τομέα της ενέργειας και στον κλάδο του ψηφιακού κόσμου, όπου καταφέραμε και η συνάδελφος Μαρία Γκάμπριελ έκανε τη συμφωνία για την περιαγωγή ε, η οποία είχε τελεσφόρησε ούτω ώστε να υπάρξουν σοβαρές εξοικονομήσεις στον τομέα των δεδομένων ε, για τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της διαδικασίας του Βερολίνου υποσχεθήκαμε ε, έως και ένα δισεκατομμύριο ευρώ διαθέσιμο για επενδύσεις σε θέματα υποδομών μέχρι το τέλος του 2020. Και στο τέλο του 2020 θα γίνει το ίδιο. Έχουμε τη συνεργασία στον τομέα τη νεολαίας ε, που εντείνεται και επίσης ε, είχαμε και την πρωτοβουλία για ε, έναν περιφερειακό οικονομικό χώρο ο οποίος οδήγησε στο ενδιάμεσο το ότι το περιφερειακό εμπόριο σε, από το 2016 και μετά αυξήθηκε κατά πολύ. Δεν αύξησε μόνο το εμπόριο μεταξύ των χωρών ε, στην περιοχή, ε, έδωσε συγκεκριμέ, και συγκεκριμένα ε, αποτελέσματα. Στην τελευταία ετήσια συνεδρίαση για τη διαδικασία του Βερολίνου στο Πόζον τον Ιούλιο ε, αποφασίσαμε και την πρωτοβουλία για μια πράσινη ατζέντα στην περιοχή. Με τα Media Days ε, δημιουργήσαμε ένα σχηματισμό ο οποίος ε, σε διάφορες επίσημες εκδηλώσεις, σε διάφορες χώρες δεν βρήκε πάντα συμφωνία για να το πω απλά αλλά είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που δημιουργεί δυνατότητες στην περιοχή αυτή εκπρόσωποι του τομέα των μέσων, όχι μόνο δημοσιογράφοι, αλλά όλοι όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα ε, και από τη Γερμανία να βοηθήσουν για μια ανεξαρτησία του τύπου και των μέσων, ε, να βελτιωθεί η κατάσταση. Έχουμε τα investments, τις επενδύσεις στην περιοχή που, για τις οποίες δώσαμε κίνητρα και το 2016 για πρώτη φορά Όλοι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων τη περιοχή και στην περιοχή, στο Σεράγεβο, σε μια, συναντήθηκαν σε μια συνάντηση εκεί. Τότε ήταν κάτι εντελώ νέο. Εμεί το θεωρούμε απολύτω φυσιολογικό όταν να συναντηθούν. Υπήρξαν πάρα πολλέ διμερεί συναντήσει μεταξύ κυβερνήσεων. Όλα αυτά τα τελευταία χρόνια τα πετύχαμε εμεί με την υποστήριξη μα. Τώρα για συγκεκριμένες ε, χώρες, ε, πιο συγκεκριμένα κάποια πράγματα τα γνωρίζετε. Για παράδειγμα η Αλβανία η οποία ε, χρειάζεται δικαστικές μεταρρυθμίσεις. όπου είναι υποδειγματικές αυτές οι μεταρρυθμίσεις για τα Δυτικά Βαλκάνια μέχρι στιγμή, στη Βοσνία Ζεγοβίνη, όπως και στο Κωσυφοπαίδιο. Έχουμε τη Συμφωνία Σύνδεσης, ε, η οποία τώρα έχει συναυθεί. Στη Φωσνία Ζεγοβίνη κατέστη δυνατό μετά από διαπραγματεύσεις να απαντηθεί το ερωτηματολόγιο μας ως προετοιμασία για τα επόμενα βήματα για μια πιθανή διαδικασία προσχώρησης. Το αναφέρω αυτό διότι ε, για να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα χρειάστηκε να στηθεί ένας ε, συντον, μηχανισμός συντονισμού εντός της χώρας με τον οποίο η χώρα κατάφερε να απαντά με μία φωνή και ήταν επιτυχές το εγχείρημα ε, και αποτέλεσε τεράστια πρόοδο στο Μαυροβούνιο όπως και στη Βόρεια Μακεδονία. Ε, στο Μαυροβούνιο έχει ήδη συναυθεί και ε, ετοιμάζεται για τη Βόρεια Μακεδονία να συναυθεί αυτό δεδομένη της ευρωπαϊκής προοπτικής και η προσχώρηση στο ΝΑΤΟ. Αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτό ότι το άνοιγμα του πρώτου κεφαλαίου πράγματι οδηγεί σε ε, διεθνή ε, πορεία. Είναι μια τεράστια, τεράστιος ο κατάλογος των επιτευγμάτων. Σίγουρα μπορεί κανείς, ε, κανείς να πει και πόσα δεν επιτέχθησαν, διότι πολλά δεν καταφέραμε να κάνουμε αυτό, είναι αδιαμφισβήτητο. Ωστόσο, συμπερασματικά, χωρίς αυτή τη, την ρεαλιστική απτή ευρωπαϊκή προοπτική, δεν θα είχε επιτευχθεί σχεδόν τίποτα από όσα μόλις σας είπα. Δεν θα είχε καταστεί τίποτα δυνατόν. Και τώρα βλέπουμε τις πρώτες αντιδράσεις. Ε, λόγω αυτή τη μη επίτευξη του να δοθεί το πράσινο φω ε, για τι διαπραγματεύσει ε, Βορεια Μακεδονία και Αλβανία, πόσο πολύ η μόχλευσή μα έχει υπονομευθεί τώρα στην περιοχή όσον αφορά τα επόμενα βήματα, τι επόμενε μεταρρυθμίσει που θα μπορούσαν να είχαν γίνει. Για το διάλογο που θα γινόταν ε, όπως και με το κοσυφοπαίδιο, να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις. Ε, το να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση στη Βοσνία Ριζεγοβίνη, αυτό θα επηρεαστεί και από αυτή τη μία απόφαση. Και ελπίζω το λάθος αυτό που διεθνώς ε, αμάβρωσε την εικόνα μας να το αποκαταστήσουμε στο μέλλον, ούτω ώστε να μην καταλήξει να είναι ένα ιστορικό σφάλμα. Ανέκαθεν έλεγα και επιμένω ότι όλοι όσοι έχουν την άποψη ότι χρειάζεται για την επόμενη διεύρυνση ε, αναθεώρηση των εσωτερικών μας κανόνων και των εσωτερικών μας διαδικασιών, πώς λαμβάνουμε αποφάσεις κτλ. Όλα αυτά είναι σωστά. Και τα δύο αυτά πρέπει να γίνονται όμως παράλληλα. Διότι αν κάνω μόνο το ένα από αυτά, δηλαδή μόνο τις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις, και μετά μόλις γίνουν οι μεταρρυθμίσεις, τότε ασχολούμαι με το ζήτημα της πιθανής ε, διεύρυνσης. Μέχρι τότε αυτές οι χώρες, ε, η προοπτική τους ε, θα πάει στη δεκαετία του 30 και δεν δίνουμε μία αξιόπιστη εικόνα ότι αυτή η προοπτική είναι αξιόπιστη. Όσον αφορά την αξιοπιστία, και αυτό είναι κάτι το οποίο ε, αμαυρώθηκε. Η Ευρώπη, όπου, η οποία παγκοσμίω ε, αγωνίζεται ε, και ισχυρίζεται ότι επιτυγχάνει πολυμερείς επιτυχίες ε, σε υψηλό επίπεδο, εμείς με αυτή την μη απόφαση σε αυτό το κλάδο έχουμε υποστεί πλήγμα, διότι η αξιοπιστία μας επλήγει. Ένα από τα μεγαλύτερα ατού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι υποσχέσεις που κάναμε ότι όταν θα πληρούνται τα κριτήρια ή σε κάποιο βαθμό τέλο πάντων την υποσχέση αυτή δεν την τηρήσαμε και ελπίζω ότι θα διορθώσουμε την εικόνα αυτή η οποία πλήγει. Σημειώστε η μεγάλη συντριπτική πλουσία των κρατών μελών ε, είναι της ίδιας άποψης πιστεύω εδώ και χρόνια ε, να ξανανοίξουν δηλαδή οι διαπραγματεύσεις. Έτσι έχουν τα πράγματα. Θα πρέπει να προσέξουμε να μην υπάρξει κάποιο κενό, διότι οποιοδήποτε κενό θα πρέπει να συμπληρωθεί αργά ή γρήγορα και πρέπει να προσέξουμε το πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Εγώ πιστεύω ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουμε τις αντίστοιχες δια, δια, συζητήσεις ε, και τους διαλόγους με τα εν λόγω κρατημέλη. Ανεξάρτητα από αυτό πιστεύω ότι είναι σημαντικό να βοηθήσουμε την οικονομική ανάπτυξη της ε, περιοχής ε, με πολύ απτό τρόπο, διότι η οικονομική ανάπτυξη θα οδηγεί σε κράτος δικαίου. Και αυτοί είναι οι δύο στόχοι που θέλουμε, το κράτος δικαίου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την οικονομική ανάπτυξη. Αυτή είναι η στόχη μας. Ε, ε, ε, οι διαδικασίες που ακολουθούμε στην Ανατολική Γειτονία, ξέρετε ότι φέτος ε, έχουμε 10 χρόνια πολιτική γειτονία. Πιστεύω ότι στην αρχή δεν ήταν πολύ καθαρό προς ποια κατεύθυνση κινούμασταν. με τον καθορισμό των 20 deliverables μέχρι το 2020 πιστεύω εκεί δόθηκε ένα σαφές περιεχόμενο, μια σαφής κατεύθυνση την οποία βλέπαν θετικά και οι εταίροι μας και την εφάρμοζαν. Και τώρα ε, κάνουμε προσπάθειες ε, για την περαιτέρω εκπόνηση της επόμενης γενιάς αυτών των deliverables μέχρι το 2030 ούτω ώστε να εφαρμοστούν αυτά ομαλά από τη μία γενιά στην επόμενη. Στι επιμέρου χώρε πολλά πράγματα, κάποια πράγματα είναι ήδη έτοιμα. Ε, και όπου υπάρχουν ερωτήσει για τι αντίστοιχε ε, χώρε, μπορούμε να τι αναλύσουμε. Στη νότια γειτονία η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική. Αρκετά διαφορετική. Ενώ στην ανατολική γειτονία ε, έχουμε την ανοικοδόμηση ως σκέψη, ως πρώτη σκέψη στον Νότο ε, είναι περισσότερο θέμα διαχείριση κρίσεων, η διαχείριση κρίσεων το βασικό θέμα. Ε, και σε καθημερινή βάση παρακολουθείτε και εσείς φαντάζομαι την κατάσταση από τη Συρία μέχρι το Μαρόκο. Υπάρχουν ε, καλές και κακές στιγμές. Εγώ ήθελα εδώ, αν μη τι άλλο, να καταφέρουμε να αναπτύξουμε λίγο περισσότερη σταθερότητα στην επόμενη ατζέντα, πιστεύω, ε, στο επόμενο σημείο τη ατζέντα θα μιλήσουμε για το Μαρόκο, αλλά αν δούμε και την κατάσταση στην Τινησία, βλέπουμε πόσο ευ, εύθραυστη είναι η δημοκρατική δομή σε αυτές τις αραβικές χώρες. Ε. Οπότε και στο μέλλον θα πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε και εδώ να παρέχουμε την υποστήριξή μας. Αυτά είχα να πω εν συντομία. Ε, για την τρέχουσα κατάσταση στη γειτονία μας ε, στα Δυτικά Βαλκάνια. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ αγαπητέ Επίτροπε. Μάθαμε κάποια πράγματα για το ιστορικό, τις επιτυχίες ε, της πολιτικής γειτονίας τα τελευταία πέντε χρόνια, αλλά και τα προβλήματα και τις απογοητεύσεις που είχαμε ειδικά αυτά τα οποία είπατε για Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία τα οποία συμφωνούν οι περισσότεροι συνάδελφοι. Να δώσω κάποιες πληροφορίες. Η συνάντηση των συντονιστών έλαβε χώρα χτες και ε, έλαβαν πολλές σημαντικές αποφάσεις. Ε, εν μεταξύ Έχουν συναντηθεί όλοι οι αρμόδιοι σκιώδεις ε, εισηγητές ε, και εισηγητές για τα Δυτικά Βαλκάνια και είπαμε ότι θα έχουμε τέσσερις ομάδες εργασίας. Μία για τα Δυτικά Βαλκάνια, μία για την Ανατολική Γειτονία, μία για την Νότια Γειτονία και μία για τα ε, χρηματοοικονομικά μέσα. Αυτά όσον αφορά τις δομές. Αν συμφωνείτε δεν χρειάζεται να αφιερώσουμε πολύ χρόνο στο Μαρόκο. Έχουμε 30-35 λεπτά για μια συζήτηση. Γνωρίζω πως πάρα πολλοί συνάδελφοι μου ζητήσει το λόγο. Άρα προτείνω να δώσουμε δύο λεπτά στον κάθε ομιλητή για να έχει μετά την ευκαιρία και ο κύριος Χάν για να απαντήσει. Ξεκινάμε ο συνήθως από τις ομάδες. Για το ΕΛΚ η κυρία Κανιέτε. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον Επίτροπο για την εξαιρετικά καλή συνεργασία που έχουμε. Σωμάδα του ΕΛΚΑ με το γραφείο σας. Εγώ πραγματικά έχω συγκινηθεί γιατί η δική μου η ευθύνη, ο τομέας αρμοδιότητας ήταν οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και πραγματικά ντρέπομαι όταν θυμάμαι που συναντούσα τον πρέσβη τη Βόρεια Μακεδονίας και του έλεγα λύστε το θέμα και έχετε μπει. Αυτό ε, το είχα υποσχεθεί πολλές φορές και εσείς το είχατε πει και πολλοί από εμάς. Δηλαδή το, το πλήγμα στην αξιοπιστία της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τεράστιο. Το σημαντικότερο τώρα είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να προχωρήσει η διαδικασία. Γιατί να έχουμε πάλι άλλη μία σύνοδο κορυφής όπου θα έχουν φρούδες ελπίδες ε, η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία θα είναι καταστροφή. Λοιπόν, όταν έγινε η Σύνοδος των ε, όταν θα γίνει η Σύνοδος των Δυτικών Βαλκανίων στην Κροατία, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να λάβουμε απόφαση. Αυτό χρειάζεται η Ευρώπη και έχει σημασία για το μέλλον της περιοχής και για την επιρροή της Ευρώπης στην περιοχή αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Καλνιέτε. Τον Νίνο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα για την ανασκόπηση της προηγούμενης θητείας που ξεκίνησε εντατικά. Βεβαίως, ναι, όλοι γνωρίζουμε τα γεγονότα της περίφημης αυτής πρότασης ότι δεν θα διευρυνθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτήν την θητεία, αλλά πολύ λίγοι μπορούσαν να προβλέψουν ότι κάποιοι βουλευτές θα ψήφισαν να φύγουν. Βεβαίω, ε, προσπαθήσαμε να το αντιμετωπίσουμε μια στρατηγική διεύρυνση. Όμως ε, έδειξε η Σύνοδος Κορυφής της Σόφιας ότι δεν συμφωνούν όλοι με αυτό. Οι εταίροι μας όμως στα Δυτικά Βαλκάνια είχαν πάρα πολύ, ε, πάρα πολύ μεγάλο ποστό της αξιοπιστίας τους το οποίο διακύβευόταν με τις χώρες αυτές αλλά και το κοσφοπόδιο για μια συμφωνία απελευθέρωσης της βίζας δυστυχώς χωρίς αποτελέσματα. Η κορατική Προεδρία χαιρέτησε τη διεύρυνση και είπε ότι είναι μία από τις προτεραιότητες της. Ελπίζω λοιπόν να έχουμε πιο θετικά αποτελέσματα στην επόμενη σύνοδο κορυφής ε, την άνοιξη στο Ζάγκρεπ. Συμφωνώ Πλήρω, ε, κύριε Επίτροπε με την ε, δήλωσή σα ότι εάν δεν εξάγουμε σταθερότητα στην περιοχή αυτή θα εισάγουμε αστάδια, αστάθεια. Με βάση λοιπόν την εμπειρία σας, ποιο είναι το μέλλον σας, ποιο είναι, με συγχωρείτε, το όραμά σας για το μέλλον. Θα αναπτυχθεί μια νέα μεθοδολογία διεύρυνσης η μεθοδολογία αυτή θα ισχύσει και για τις υποψήφιες χώρες ε, που ήδη κάνουν διαπραγματεύσεις όπως η Σερβία και το Μαυροβούνιο. Και τέλος, ποιε ε, θεωρείτε ότι θα είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις στο μέλλον. Ευχαριστώ τον Νίνο για το Ρινιού Ναταλή Αζώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ντουάζο, ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε για αυτή την ε, μακρά περιγραφή της ε, διαδικασίας διεύρυνσης. Από πλευρά μου θα σας ρωτήσω το εξής. Πρώτα-πρώτα καλή επιτυχία, αλλά δυστυχώς υπάρχουν και κάποια τα οποία συμβαίνουν που είναι λιγότερο ευχάριστα για τη Σερβία. Θέλω να σας ρωτήσω μια που την αναφέρατε. Είπατε ότι ξεκίνησε τη διαδρομή της ένταξης και έχουμε σχετικά κεφάλαια. Πέστε μας εσείς πώς το αξιολογείτε. Έχουμε αρχίσει διαπραγματεύσει με την χώρα. Τι γίνεται, υπεχώρησε η επιρροή της Ρωσίας και ο διάλογος με το Κόσοβο βελτιώθηκε και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των ε, μειονοτήτων, το κράτος δικαίου, τα πάνε καλύτερα. Άρα τι θα γίνει, τι μπορεί να γίνει και τι θα γίνει με όλες αυτές τις εξελίξεις, με αυτές τις μεταρρυθμίσεις που θέλουμε και ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να υποστρίξουμε την διεύρυνση προς τα εκεί. Θα πρέπει σίγουρα να αναθεωρηθεί η διαδικασία της προσχώρησης και συμφωνώ μαζί σας και σας ερωτώ πότε η Επιτροπή θα κάνει τη σχετική πρόταση. Υπάρχει συνένεση γιατί σήμερα τα πράγματα δεν είναι τόσο ικανοποιητικά στη συνέχεια. Πέστε μας λίγο περισσότερα σε σχέση με την εταιρική σχέση με την Νότια Μεσόγειο. Σα είπατε ότι είναι σε κατάσταση κρίση. Τι γίνεται με την Τινησία. Θα πρέπει στο μέλλον να υποστηριχθεί η χώρα. Ε, είπατε, μου φαίνεται ότι αυτό είναι πάρα πολύ σύντομο ως δήλωση γιατί το μέλλον για το Μαγκρέμπ, για την Νότια Μεσόγειο, ε, για τη δημοκρατική παράδοση της Τινησίας, όλα αυτά έχουν σχέση με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το επηρεάζουν. Οπότε πραγματικά θα πρέπει με αυτή την ε, ευκαιρία εδώ να μας πείτε εις βάθος τι γίνεται, τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο για να βοηθήσουμε την Τινησία. Ευχαριστούμε. Βιόλα το Μπάτλ. Σε ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, κύριε Χάν. Αναφέρατε διάφορα ζητήματα, το πλήγμα στην αξιοπιστία, ότι είναι πολύ σημαντικό να στηρίξουμε την περιφερειακή ανάπτυξη. Και Βεβαίω ήδη οι συναδελφοί αναφέρθηκαν ε, στο θέμα Σερβίας Κοσφοπεδίου και πώς μπορεί να επιτευχθεί μια επιτάχυνση του διαλόγου αυτού. Θα ήθελα επίσης ε, τις εκτιμήσεις σας για το σε ποιο βαθμό βλέπετε μια διάθεση για επιτάχυνση από πλευράς ε, Σερβίας ή Κοσοβάρων ως ε, παρατηρήτρια των εκλογών στο Κοσμοπέδιο άκουγα συνέχεια ότι ε, σε πολλά σημεία ήμασταν πολύ ήπιοι με τα εσωτερικά του κοσφοπεδίου, δεν κάναμε τίποτα για την διαφθορά, δεν ασχολούμαστε καθόλου με το κράτος δικαίου. Επίσης το ότι έχει υπάρξει μια κατάληψη του κράτους από τις ελίτ ε, την οποία δεν έχουμε αντιμετωπίσει. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλοί, είπα, Κατάρ, ε, Κίνα και λοιποί, οπότε υπάρχει μεγάλη πίεση για να μην χάσουμε την επιρροή μας, αλλά θα ήθελα να ακούσω την δική σας εκτίμηση. Χτες συναντηθήκαμε με Σέρβους ε, βουλευτές και ήμουν ε, πραγματικά δοκίμασα μια πολύ θετική έκπληξη για το πόσο δυτικοί ε, εμφανίστηκαν και πόσο θέλουν να ενταχθούν. Έχουν λάβει πρόσκληση και για το ΝΑΤΟ, αλλά μας ζήτησαν ακριβώς να αντιδράσουμε ένεργα στην ρωσική προπαγάνδα. Δηλαδή αυτό ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει λοιπόν κάποιο πρόγραμμα από πλευράς ε, κομισιών ε, για το πώς θα μπορέσουμε να ε, φέρουμε τη Σερβία πιο κοντά σε μας. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφε. Οι άλλες πολιτικές ομάδες δεν ζήτησαν το λόγο. Αιντι, ναι, ζητήσατε. Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σα άκουσα πολλέ φορέ να μιλάτε για ιστορικό λάθο. Αυτή είναι η δική σα εκτίμηση και δικαίωμα έχετε να την έχετε. Ωστόσο, δεν πρέπει να είναι γεγονό ότι έτσι λειτουργούν τα θεσμικά όργανα αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εγώ, εκ μέρου τη ομάδα μου, χαίρομαι που μερικέ φορέ αυτή η λειτουργία μα υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και μια ένωση κυρίαρχων κρατών. Τα οποία κατά καιρού μπορούν να πούν και όχι για ορισμένα θέματα. Μπορούν ε, σε ορισμένα θέματα να επιβάλλουν ε, τον κανόνα της ομοφωνίας. Η θέση της Γαλλίας ε, για το θέμα των Βαλκανίων την αναφέρατε. Εγώ χαίρομαι που η θέση του υπερασπίζει ο κύριος Μακρόν είναι αυτή που υπερασπίζεται το Rassemblement Νασιονάλ, δηλαδή λειτουργία των θεσμών και αφενός ότι κάποια στιγμή χρειαζόταν να γίνει και η συζήτηση του μέχρι πού εκτείνεται η Ευρώπη. Τι θα γίνει, θα τη διευρύνουμε διαρκώς χωρίς ε, ποτέ να ορίζουμε, να θέτουμε κάποιο όριο. Έχω τέσσερις ε, ερωτήσεις να σας κάνω. Για την Τουρκία, μέχρι πότε θα επιμένουμε να συνεχίζουμε αυτές ε, τις διαπραγματεύσεις και να... γιατί δεν κλείνουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις οριστικά. Το πραξικόπημα το ανεχτήκαμε όπως δεν έχουμε κάνει πουθενά αλλού, Την εκβιασμό για το μεταναστευτικό ζήτημα, την επίθεση κατά των Κούρδων, την ανεχτήκαμε και κάθε φορά συνεχίζουμε, λες και δεν έγινε τίποτα να διαπραγματευόμαστε. Για το κοσφοπέδιο απαιτήσατε για το πρώτο κεφάλαιο διαπραγματεύσεων όπως και με τη, η Σερβία να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του κοσφοπεδίου. Πέντε κράτη-μέλη δεν την αναγνωρίζουν. Για ποιο λόγο ορίζουμε τέτοια υποχρέωση για τη Σερβία που δεν απαιτούμε για άλλα κράτη. Εξ ονόματος πιανού και τελευταίο σημείο για το κοσφοπέδιο επίσης τέλος. Ίσως να μου διέφυγε, δεν άκουσα να καταδικάζεται ε, τις ε, ε, κυβερνητικές δυνάμεις του Κωσυφοπεδίου που μπήκαν σε θύλακες της Σερβίας και κατά πόσο υπάρχει μια σχετική απέτηση για να μπορέσει να, υπάρξει, να είναι υποψήφια χώρα του Κωσυφοπέδιου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μαριάννη. Θα ήθελα πάρα πολύ να σχολιάσω. Πάρα πολύ. Αλλά θα σιωπήσω. Απλά είμαι πρόεδρο σήμερα. Είναι πάρα πολλά πράγματα που θα ήθελα να σχολιάσω. Το ECR δεν είναι παρόν αυτή τη στιγμή. Γκουε θέλει να πει κάτι. κάποιο Όχι. Πάμε στο δεύτερο γύρο λοιπόν για το Έλκο Michael Galler. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και για τη δουλειά σας μέχρι στιγμή. Εύχομαι ό,τι καλύτερο στην καινούργια σας, στο καινούργιο σας λειτουργήμα. Συμφωνώ με την εκτίμησή σας για τα Δυτικά Βαλκάνια. Αυτές τις χώρες φυσικά μπορούμε να τις βοηθήσουμε και ενεργά γιατί τις θέλουν πολύ και ο Πούτιν και ο Ερντογάν. Δεν θέλουμε λοιπόν να γίνει κάτι τέτοιο και εγώ είμαι υπέρ επίση, οι θεσμικές ε, μεταρρυθμίσεις να γίνουν παράλληλα. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, να γίνουν και τα δύο ταυτόχρονα. Και εμεί ε, ξέρουμε ότι όταν ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσει το 2005 με την Κροατία, μετά από 8 χρόνια ε, κατάφερε η χώρα να, να μπει. Οπότε δεν γίνεται αυτό από τη μια μέρα στην άλλη. Ε, χρειάζεται μεγάλη δουλειά. Οπότε ίδια εκτίμηση έχω με εσά. Έχω μία ερώτηση για την Ανατολική Γειτονία. Ξέρετε ότι ε, εντό των έξι χωρών της Ανατολικής Γειτονίας τρει έχουν φιλόδοξη ατζέντα μαζί μα. Η Ουκρανία, η Γεωργία και η Μολδαβία. Και η ερώτησή μου, σε ποιο βαθμό θα μπορούσαμε ε, σταδιακά κάποια προγράμματα που ήδη υπάρχουν εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση να τα χρησιμοποιούμε και σε αυτέ τι χώρε, ε, να τα υιοθετήσουν και αυτέ και κατά πόσο αυτό θα ήταν υποφελέ για αυτέ. Ε, ένα προσφυλέ θέμα είναι. Δεν θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να καταργήσουμε το τέλη περιαγωγής για αυτές τις χώρες, στέλνοντας ένα μήνυμα ότι ε, να, ας πούμε κάτι μπορεί να είναι υποφελέ και για τις δύο πλευρές ε, και για τους χρήστε σίγουρα. Σα ευχαριστώ πολύ και σα εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε κύριε Γκάλερ για του σοσιαλιστές. Ε, ο κύριος Αρακόβατς, αν το είπα σωστά. Thank you, Mr. President, Mr. Commissioner. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Παρουσία δύο δικτατόρων του κυρίου Ερντογάν και του κυρίου Αλίεφ, ο κύριος Όρμπαν δήλωσε αν καταφέρουμε να πάρουμε αυτό το χαρτοφυλάκιο διεύρυνσης και γειτονίας θα είμαστε στην υπηρεσία σας για να επιτύχετε τους σκοπούς σας. Το ερώτημά μου αφορά την πολιτική γειτονίας και το σχετικό χαρτοφυλάκιο. Θεωρείτε ότι πρέπει να το λάβει η κυβέρνηση Όρμπαν ενώ εντωμεταξύ ε, συνεισφέρει στην ε, τουρκική επιθετικότητα στην Βόρεια Συρία. Ευχαριστώ κάποιες από τις ερωτήσεις αυτές ίσως να τεθούν ε, στον υποψήφιο όταν γίνει η ακρόαση. Δεν νομίζω ότι ο Γιωχάνες Χάν είναι υπεύθυνο για την ουγγρική πολιτική, αλλά εν πάση περιπτώσει ευχαριστώ. Περνάμε στον κύριο Κιουτσούκ τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που ήρθατε και απαντήσατε τις ερωτήσεις μας κύριε Επιτροπέ. Παρά την τεράστια πλειοψηφία των κρατών μελών, για τρίτη φορά σε 16 μήνες το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν συμφώνησε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει με Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία. Μετά από την απόφαση του Συμβουλίου είπατε ότι δεν πρέπει να κατηγορούμε κάποιον. Αλλά δεν ήταν και μια στιγμή δόξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμφωνούμε. Οποιαδήποτε αναβολή θα βλάψει την ε, αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωση στο Βαλκάνια και θα πρέπει να επανεξεταστεί αυτή η απόφαση ω το των δυνατών. Απ' την άλλη όμως ε, υπάρχουν ε, ακριβώ αυτά τα οποία είπατε, ότι θα πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσει. Βεβαίως δεν είμαστε ενάντια, αλλά το θέμα είναι ποιοι είναι οι όροι, ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα ή εάν αυτό θα πηγαίνει χέρι-χέρι με την διαδικασία που έχει ξεκινήσει για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Μπορείτε να επεκταθείτε λίγο. Σας ευχαριστώ κύριε Κιουτσούκ για τους ε, πράσινους κυρία Τρίκ. Ε, ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Χάν για τη δουλειά που έχει κάνει στην πολιτική διεύρυνση. Ε, τα όσα είπατε για την μία απόφαση του Συμβουλίου. Πράγματι η απόφαση αυτή ήταν ένα πλήγμα για τους πολίτες και τους πολιτικούς της χώρες ε, αυτές και βεβαίω ε, υπάρχουν και δυσκολίες το τι σημαίνει δηλαδή για τις ξένες επιρροές και τη σταθερότητα στην περιοχή και εγώ σκέφτομαι τι μπορούμε να κάνουμε μεταξύ μέχρι να ληφθεί μια νέα απόφαση για να διατηρηθεί ένα θετικό πνεύμα και ε, να υπάρξει κάποια εμπιστοσύνη και να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να συνεχίσουν τις ε, μεταρρυθμίσεις ε, για να τους στηρίξουμε. Ξέρω ότι θα γίνουν νέες εκλογές στην Βόρεια Μακεδονία. Ποια είναι η δική σας η άποψη για τον αντίκτυπο που θα έχει αυτό για την επόμενη περίοδο. Βλέπετε έχει αντίκτυπο σε, νέες, ε, σε περιοχές ή άλλες χώρες. Και ξέρετε βεβαίως ότι είχαν πολλές συζητήσεις και διαφορετικές απόψεις ε, για την διασύνδεση μεταξύ Βόρειας Αλβανία, Μακεδονίας και Βόρειας Αλβανίας. Ε, ποια είναι η άποψή σας τώρα για την απόφαση του Συμβουλίου να μην ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις. Συζητιέται αυτό καθόλου. Ευχαριστώ κυρία Στρίκ. Τρίτος γύρος. Για το ΕΛΚ, ο κύριος Καμπυλίους. Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, και εγώ να σας ευχαριστήσω. Είναι το έργο που επιτελέσατε απίστευτο. Βεβαίω και πάντοτε θέλουμε να σημαίνονται πρόεδρο στην υπόθεση της διεύρυνσης. Βέβαια, είχατε αναλάβει τον προϋπολογισμό ε, για τα σχετικά και δεν θα τα ξεχάσετε. Θα κοιτάτε και προς εκείνη την κατεύθυνση, αλλά ξέρετε την περίφημη ρίση ότι αντί να εισάγεται αστάθεια θα πρέπει να εξάγετε σταθερότητα. Πώς μπορείτε εσείς να το πετύχετε αυτό στην γειτονιά μας σε σχέση με την διεύρυνση. Είδαμε την τελευταία απόφαση του Συμβουλίου και μπορούμε να πούμε ότι η πολιτική διεύρυνση βρίσκεται σε κρίση. Οπότε από τη μια μεριά, από τη μια μεριά μπορεί κανεί να αγωνία για το τι θα γίνει. Αλλά αν κανεί ρίξει μια ματιά στην ιστορία, θα διαπιστώσει ότι από τι κρίσει πάντα βγαίνει κάτι καλό. Ότως ώστε με κάποια διαβήματα να γίνει αποτελεσματική και πετυχημένη η πολιτική αυτή. Οπότε πέστε μας λίγο περισσότερα, τι θα προτείνετε. Ε, τι θα λέγατε στους ε, διαδόχους στην Επιτροπή, πώς θα έπρεπε να οργανωθούν για να αποφύγουμε τέτοια πράγματα που να μπλοκάρει μια χώρα το προτσές. Επίσης, για πέστε μας. Μας ε, η πολιτική εταιρική σχέση είναι πολύ σημαντική και ο Μικαλ Γκάλερ σας ανέφερε και σας ερώτησε τι μπορείτε να κάνετε για να υπάρξει κάποια διαφοροποίηση μεταξύ των έξι αυτών χωρών που άλλες πάνε καλύτερα, άλλες λιγότερο καλύτερα. Οπότε, μια στρατηγική για Μολδαβία, Γεωργία, Ουκρανία, αυτές οι χώρες να μπορέσουν να τα πάνε καλύτερα. Ο Πρόεδρος, κυρία Σάντος, για τους Σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα-πρώτα, συγχαρητήρια, κύριε Επίτροπε, για τα όσα κάνετε και όσα κάνατε και τις καλύτερες ευχές μας για το μέλλον. Για πέστε μας λίγο περισσότερα για τις αποφάσεις ή τις μη αποφάσεις του Συμβουλίου γιατί είχαν δημιουργηθεί κάποιες αυξημένες προσδοκίες για Αλβανία και Σκόπια. Είχαμε όλη αυτή τη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων, είχαμε τον διάλογο, στη συνέχεια ε, είχαμε περισσότερες προσπάθειες και εσείς μας αναφέρατε για τις επενδύσεις τόσων ετών από ό,τι φαίνεται. Το αποτέλεσμα δεν ήταν και τόσο τρομερό. Καταλήξαμε τώρα να έχει υποστεί με εμπιστοσύνη του κόσμου στις ώρες εκείνες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για πετε μας, πώς θα βγείτε από το αδιέξοδο, τι θα κάνετε, τι θα πείτε στον κόσμο αυτό. Κάνανε τις μεταρρυθμίσεις. Ήταν επώδυνε κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, για την κοινωνική συνοχή. Και θα ήθελα να με βοηθήσετε να καταλάβω οι προθέσεις μας άλλαξαν. Θέλουμε να συνεχίσουμε τη διαδικασία αυτή Θέλουμε μήπως να βοηθήσουμε τη μία χώρα στην προσχώρηση και άλλη να μείνει στο θάλαμο αναμονής. Γιατί υπάρχουν δείξει ότι πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν θα πρέπει να έχει κενά η πολιτική. Θα πρέπει κάτι να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλιώ άλλο θα έρθει να γεμίσει αυτό το κενό. Ο πρόεδρο, σα ευχαριστώ. Renew. Γκέτα. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για όσα μας είπατε για τη συμβολή στη συζήτησή μας και επιτρέψτε μου την εξής παρατήρηση. Παρατήρηση υπομορφή ερωτήσεως. Είναι δυνατόν τα θέματα της διεύρυνσης της Ένωσης να φύγονται χωρίς να φύγεται το άλλο θέμα το πολύ πιο σημαντικό και πιο δραματικό το θέμα της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι εδώ ξέρουμε ότι η Βόρεια Μακεδονία και ίσως η Αλβανία έχουν ενδεχομένω εσωτερικές ε, δυσκολίες, εσωτερικά προβλήματα λόγω των προσφάτων αποφάσεών μας. Γνωρίζουμε την πολιτική δυσκολία, το στρίμωγμα αυτό που έχει γίνει σε διάφορες πρωτεύουσες, ε, Ρώμη, Βερολίνο και Παρίσι, έτσι ενδεικτικά σας τις αναφέρω αυτές. Άρα, είναι δυνατόν να ασχολείται κανείς με την διεύρυνση χωρίς να ασχολείται με την κατάσταση της Ένωσης. Ευχαριστώ. Και εμεί ευχαριστούμε λοιπόν. Τώρα έχουμε άλλου τέσσερι αγορητέ. Ε, να είσαστε όσο ε, γίνεται πιο σύντομοι για να μιλήσουν όλοι. Και μετά να έχει 10-15 λεπτά ο κύριο Χάν για να απαντήσει. Αλεξάνδροφ, ο επόμενο. Ευχαριστούμε, κύριε. Επίτροπε. παρακολούθησα τις προσπαθίες σας σε σχέση με τη Βόρεια Μακεδονία και σήμερα μπορώ να διαβεβαιώσω όλους ότι με άριστο τρόπο εκπροσωπήσατε εκεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βοηθήσατε την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης στην Βόρεια Μακεδονία. Την εμπιστοσύνη έναντι του Ευρωπαϊκού Ιδιώδους. Και σε σχέση με αυτά που άκουσα από τους συναδέλφους μπορώ να πω το εξή. Εάν δεν αναλαμβάνει η δράση Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλος το κάνει αυτό. Η Ρωσία και η ιστορία είναι μάρτυρας τούτου. Ήδη έχει ξεκινήσει αντιευρωπαϊκή πολιτική και πολιτική κατά του ΝΑΤΟ εκεί. Η σερβική κυβέρνηση και η ηγεσία της χώρας ισχυρίζονται ότι η Σερβία είναι κάτι σαν δορυφόρος της Ρωσίας στα Βαλκάνια. Θωρακίζονται οικονομικά, θωρακίζονται όσον αφορά τη συνεργασία τους με την Ρωσία. Πρόκειται για τα ευρωπαϊκά σύνορα οι θεμελιώδεις ελευθερίες και τα δικαιώματα ε, πρέπει να γίνονται σεβαστά και το κράτος δικαίου. Η, η Ρωσία είναι εκτός των συνόρων παρά ε, την φιλία Ρωσίας-Γαλλίας. Βόρεια Μακεδονία, Μαυρό Βούνιο και ελπίζουμε η Σερβία αλλά και το Κωσυφοπαίδιο θα πασχίσουν να πετύχουν τις ευρωπαϊκές ε, αξίες. Η δε Βουλγαρία έχει διατρονώσει την άποψή τη ότι υποστηρίζει τη διεύρυνση προ τα εκεί, δηλαδή για Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία. Και τώρα για τους σοσιαλδημοκράτες η κυρία Αρενά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με την Αταλή Λουαζό. Υπάρχει ανησυχία για ε, αισθάνομαι κάποια ανησυχία γιατί δεν συζητήσαμε για την νότια εταιρική σχέση. Ξέρετε, στο Κοινοβούλιο ψηφίσαμε, είχαμε ένα ψήφισμα όσον αφορά την κατάσταση στην Αίγυπτο, σημαντικό εταίρο στη Μέση Ανατολή και στο Μαγκρέμπ ε, ειδικότερα. Έχω λοιπόν δύο ερωτήσεις. Πρώτον, έχουν παγώσει κάποιες συνεργασίες με την Αίγυπτο. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα έχει ξεπαγώσει ή έχει ξαναμπλοκάρει η κατάσταση από την Κομισιόν όσον αφορά τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων δράσεων και τι μέτρα έχει υιοθετήσει η Κομισιόν ε, λόγω του ότι η Αίγυπτος ε, προφανώς δεν σέβεται το εμπάργκο όπλων προς τη Λιβύη. Τι γίνεται ε, από αυτήν την άψη στην Κομισιόν. Ευχαριστούμε Μαρία, κύριε Μουτσέβιτς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε και, ε, κύριε Επιτροπέ να σας δείξω κάτι. Κοιτάξτε, να σας δείξω αυτό. Αυτή η τσάντα την πήρα το 2003 στη Θεσσαλονίκη και την κουβαλάω μαζί μου γιατί έτσι εκφράζω προσωπικά την ελπίδα ότι η υπόσχεση που έγινε από, την κυρίαρχη, από τα κυρίαρχα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι τα κράτη των Βαλκανίων θα ενταχθούν στην Ένωση θα εκπληρωθεί, να δείξουμε το σεβασμό μας για αυτούς. Αλλά αφού είστε αρμόδιος και για τη γειτονία, θα σας ρωτήσω για έναν από τους ανατολικούς μας εταίρους. Εγώ ζω σε ένα σπίτι το οποίο είναι δύο χιλιόμετρα από το σύνορο με τη Λευκορωσία. Τι θα κάνετε με τη Λευκορωσία που είναι μια δύσκολη γείτονα χώρα. Thank you, and finally, Mr. Mavridis. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μαυρίδης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην προηγούμενη θητεία υπήρξαν αρκετές φορές που διαφώνησα μαζί σας και υπήρξαν και αρκετές απογοητεύσεις. Τώρα επειδή ίσως να είναι και τελευταία φορά που έχουμε αυτή τη συνάντηση με την ιδιότητά σας για τα θέματα ε, ε, enlargement, θα σας πω κάτι που το θυμάμαι χαρακτηριστικά και είναι μια τολμηρή δήλωσή σας σε μια καθοριστική στιγμή ειλικρίνειας. Δεν θα ξεχάσω όταν διερωτηθήκατε, όπως και όλοι μας, όταν έγινε το πραξικόπημα στην Τουρκία, πώς βρέθηκαν ξαφνικά εκείνες οι δεκάδες χιλιάδες ονόματα σε καταλόγους τα οποία ο Ερτογάν είχε έτοιμα για να κυνηγήσει. Ε, προφανώς όλοι γνωρίζουμε τι είχε συμβεί. Τώρα έρχομαι σε κάτι άλλο όμως που θέλω την άποψή σας. Είναι μια περίεργη κατάσταση με την Τουρκία. Αφενός επίσημα είναι υποψήφια για ένταξη χώρα και ταυτοχρόνως θα σας πω δύο καταστάσεις. Πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάνθηκε ότι η συμπεριφορά της είναι έκδηλα παράνομη σε τέτοιο βαθμό στην Ανατολική Μεσόγειο και στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας που θα πρέπει να τις επιβληθούν κυρώσεις. Τόσο έκδηλα παράνομη. Και το δεύτερο είναι ότι σε σχέση με τα Δυτικά Βαλκάνια, που όλοι θέλουμε να κινηθούμε η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση να κινηθούμε γρήγορα για να γεμίσουμε την περιοχή και να σπρώξουμε μακριά την ρωσική επιρροή, αλλά η Ρωσία δεν είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε έχουμε κάποια ιδιαίτερη σχέση, αλλά να διώξουμε και την τουρκική επιρροή. Δεν είναι περίεργο. Δηλαδή τελικά είναι επίσημη χώρα, είναι στρατηγικός εταίρος για ένταξη κλπ. Και ταυτοχρόνως ανταγωνιζόμαστε απέναντι στην τουρκική επιρροή. Θέλω να ακούσω την άποψή σας σε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πάντως για όλα όσα έχετε συνεισφέρει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις ε, συνεισφορές σας. Ε, κύριε Χάν, ακούσατε πολλά και διάφορα. Μια που έχουμε τόσες ερωτήσεις, ε, θα έλεγα να μιλήσετε 10-15 λεπτά, αλλά μόνο εάν μου υποσχεθείτε, συνάδελφοι, ότι δεν θα γίνει τόσο εκταμένη συζήτηση για το Μάρκο. Γιατί βεβαίως έχουμε και την συνάδελφο εδώ πέρα σε 15 λεπτά. Την Αντζελίνα. Κοιτάξτε. ε, για το κάθε θέμα τελικά θα έπρεπε να κάνουμε ξεχωριστή συνεδρίαση νότια γειτονία, ανατολική κτλ. Νομίζω ότι σήμερα ήταν το βασικό θέμα τα Βαλκάνια, αλλά θα αναφερθώ σε όλες τις ερωτήσεις. Για τα Δυτικά Βαλκάνια να υπενθυμίσω ακόμη μια φορά, νομίζω δεν αμφισβητεί κανείς ότι ε, αυτές οι έξι χώρες ε, οι οποίες ε, γειτονεύουν ε, με χώρες της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης έχουν σύμφωνα με το άρθρο 49 το δικαίωμα να ζητήσουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν να τα δούμε αυτά τα πράγματα σοβαρά και βεβαίω υπόθηκε από διάφορους ομιλητές πως ε, τα τελευταία χρόνια ε, ή τις δεκαετίες αν θυμηθούμε την ε, Θεσσαλονίκη υπήρχε η υπόσχεση ότι οι χώρες αυτές έχουν μια προοπτική και αυτό ακριβώς είναι το θέμα της αξιοπιστίας μας. Το εάν δηλαδή αυτά τα οποία υποσχόμαστε τα λέμε σοβαρά, ναι ή όχι και αυτή τη στιγμή πρέπει να το πούμε έχουμε ένα πρόβλημα αξιοπιστίας γιατί στο θέμα της ε, Βόρειας Μακεδονίας και Αλβανίας ε, υπήρξαν σαφείς ε, όροι και λέγαμε ότι όταν εκπληρωθούν θα μπορέσουν να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις και οι όροι αυτοί είχαν τεθεί ομόφωνα από όλα τα κράτη-μέλη. Δεν ήταν ότι η Κομισιόν αποφάσισε κάτι μόνη της και τις επέβαλε στις χώρες αυτές. Ήταν αποτέλεσμα εκτεταμένων διαπραγματεύσεων των 28 κρατών μελών με τις χώρες αυτές. Δεν ήταν κάτι το οποίο επιβλήθηκε. Ήταν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ευρύτατης. Και όταν μετά από μια τέτοια αξιολόγηση, μετά από τόσες συζητήσεις με μεγάλη διαφάνεια, ε, εκπλήρωσαν οι χώρες αυτές ε, τις ε, διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι αυτονόητο ότι θα αντιδράσουμε θετικά και θα ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις. Και Θα συμφωνήσω με αυτούς που είπαν ότι η αρχή των διαπραγματεύσεων και ε, επί τη ευκαιρία πράσινο φως δεν σημαίνει ότι ξεκινάνε αμέσως οι διαπραγματεύσεις, πρέπει να προετοιμαστούν. Δηλαδή ανάμεσα στο πράσινο φως και το άνοιγμα του πρώτου κεφαλαίου πάλι περνάνε μήνες. Και το άνοιγμα του πρώτου κεφαλαίου απαιτεί και αυτό ομόφωνη απόφαση όλων των κρατών μελών. Δηλαδή το πράσινο φως πραγματικά θα ήταν κατά κυριολεξία ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα για να ξεκινήσουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Μια αναγνώριση των μέχρι τώρα προσπαθειών. Και βεβαίω Σημασία έχει και το τι σημαίνει αυτό για τι άλλε χώρε Το είπα και θα το ξαναπώ. Είδαμε πώς ε, ολοκληρώθηκε η Συμφωνία των ε, Πρεσπών, ποιε θετικές επιπτώσεις ε, είχε στην περιοχή σε σχέση με αυτό το οποίο λέω αν θέλετε μια θετική φιλοδοξία Δηλαδή ο διάλογος ε, μεταξύ Σερβίας ε, και Κωσφοπεδίου απέκτησε νέα ενέργεια γιατί δεν ήθελα να μείνουν πίσω όταν οι άλλοι ε, είχαν τόσο καλά αποτελέσματα. Λοιπόν, επέδρασε και στις άλλες χώρες της περιοχής που δεν ήθελα να μείνουν πίσω. Λοιπόν, κάθε θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης για μία χώρα φέρνει μαζί του θετικές αντιδράσεις ε, στις άλλες χώρες. Και ακοντράριο από την άλλη, αν δεν ε, κάνουμε κάτι, υποφέρει η επιρροή μας ε, στις άλλες χώρες. Και κάνατε κάποιες ερωτήσεις για το τι γίνεται με τον διάλογο Σερβίας-Κοσφοπεδίου. Θα σας πω ανοιχτά λοιπόν ότι ε, από την ε, σερβική σκοπιά ο διάλογος αυτός έχει νόημα αν υπάρχει κάποιο θετικό αποτέλεσμα δηλαδή μια διευθέτηση μεταξύ των δύο χωρών μόνο εάν υπάρχει ευρωπαϊκή προοπτική και από την ε, πλευρά του κοσφοπεδίου όπου υπάρχουν θετικές ε, πολιτικές εξελίξεις ε, στη χώρα αυτή. Ελπίζω προσεχώς να σχηματιστεί η κυβέρνηση, η οποία θα επικεντρωθεί παραδείγματος χάρη στο έλλειμμα κράτους δικαίου. Αλλά το μεγάλο κίνητρο, το καρότο, εάν θέλετε, είναι η ευρωπαϊκή προοπτική και βεβαίως ε, δικαίως ε, μιλάμε πολύ γι' αυτό και στις ίδιες τις χώρες λένε όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις που ζητάει από μας η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι κατά κύριο λόγο πρωτίστως προς το συμφέρον των πολιτών. Δεν είναι για να χαρούμε εμείς εδώ σε αυτή την αίθουσα αλλά για να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής των ανθρώπων ε, στις χώρες αυτές. Και προφανώς εδώ πέρα η κύρια κινητήριος δύναμη είναι η ευρωπαϊκή προοπτική, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην ε, περιοχή αυτή και αυτό αφορά και τις ε, χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το λεγόμενο brain drain, το ότι οι νέοι με προσόντα με κίνητρα φεύγουν και πάνε ε, σε άλλα μέρη της Ευρώπης. Ε, κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά όχι με το στόχο να μάθουν κάτι και να επιστρέψουν. Όπως ε, το Εράσμους που θα ήταν το ιδεώδες, αλλά με το στόχο να παραμείνουν εκεί. Στην καλύτερη περίπτωση να επιστρέφουν στην οικογένεια για διακοπές και να κάνουν εμβάσματα, αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν, δεν ε, μπορεί να είναι προς το σύμφωνο μας ε, στην καρδιά της Ευρώπης, όπως ε, στα Δυτικά Βαλκάνια, που είναι εσωτερική αυλή, αν θέλετε, της Ευρώπης, να προκαλούμε να ερημώνουν ολόκληρες περιοχές από ανθρώπους και να υπάρχει κατά κυριολεξία ένα κενό και ένα κενό ασφαλείας μετά το οποίο οπωσδήποτε δεν συνεισφέρει στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Λοιπόν, μην ε, έχουμε ψευδεστήσεις. Ε, εντάξει, βλέπουν βεβαίως και μόνο τους ότι χρειάζονται αυτές οι μεταρρυθμίσεις, αλλά υπάρχει και η πίεση της ευρωπαϊκής προοπτικής, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι σε αυτές τις περιοχές το επιθυμούν και θέλουν να κάνουν αυτές τις μεταρρυθμίσεις ίσως όχι ταχύτητα που θα θέλαμε, αλλά οπωσδήποτε μόνο ε, χάρη σε αυτήν την ευρωπαϊκή ε, προοπτική. Και γι' αυτό θα έλεγα ότι χωρίς ε, αυτό, χωρίς αυτή την απλή διαπίστωση, δεν θα έχουμε επιρροή στην περιοχή, που είναι και προς το συμφέρον των ανθρώπων και προς το δικό μας και πολλά από τα ερωτήματα τα οποία θέσατε, το τι είναι σωστό, το τι είναι δυνατό για την απόφαση, τη μη λήψη απόφασης ε, ε, για όλες τις χώρες ουσιαστικά πλην του Μαυροβουνίου έχουμε συνομιλήσει. Επίσης, παρατηρούμε ότι πλέον ε, έχει χαθεί η ορμή, αν θέλετε, η δυναμική και δεν είναι εύκολο να αποκατασταθεί για να κινηθούν ε, κάποια πράγματα. Ε, ρωτήσατε επίσης για τη ρωσική επιρροή. Νομίζω ότι δεν πρέπει να ξέρετε ότι η Σερβία έχει κάνει περισσότερες ασκήσεις με τον ΝΑΤΟ παρά με τη Ρωσία. Αλλά η εντύπωση η οποία υπάρχει για την Σερβία είναι ακριβώς το αντίθετο. Λοιπόν, εδώ πέρα πρέπει όλοι να συνεισφέρουν στο θέμα αυτό των ε, χωρών ε, αλλά και των χωρών αυτών αλλά και οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα λοιπόν του πώς θα προχωρήσουν περαιτέρω οι διαπραγματεύσεις έχει συζητηθεί, αλλά ε, θα σας πω ότι ε, είναι κάτι το οποίο υπάρχει δηλαδή καμία από αυτές τις διαδικασίες δεν οδηγεί αυτομάτως ε, σε ένταξη όπως ξέρετε τελικά κρίνεται η δυνατότητα ένταξης μιας χώρας ε, με την ΔΕ Τουρκία έχουμε, διαπιστώ, έχουμε πει ρητός πως το αποτέλεσμα είναι ανοιχτό, το τελικό αποτέλεσμα και ότι αν υπάρξουν υπαναχωρήσεις στο κράτος δικαίου θα πρέπει να διακοπούν οι διαπραγματεύσεις. Από την άλλη, βεβαίως πριν από λίγα χρόνια απειλήσαμε το Μαυροβούνιο, κατόπιν οδήγησε βεβαίως σε μια νέα όθηση Είχαμε λοιπόν διάφορες ε, δυνατότητες ε, για να αντιδράσουμε και προτείναμε για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο να μην ε, τα χωρίσουμε ανά χώρες, αλλά να υπάρξει μια θεματική κατανομή των χρημάτων για να είμαστε και πιο ευέλικτοι να υπάρξει και ένας ανταγωνισμός μεταξύ των ε, χώρων. Αλλά και πάλι θεωρώ ότι οι συνεργάτες μου και οπωσδήποτε η διάδεχός μου ε, θα είναι ανοιχτή. Εντάξει, κανείς δεν είναι τέλειος, μπορούν να τα ξαναδούν αυτά τα πράγματα, αλλά είναι σημαντικό να γνωρίζουμε εάν τα λέμε σοβαρά ή εάν ε, ήταν απλά Κάτι το οποίο λέγαμε για να πούμε τελικά δεν μπορούν να ανοίξουν διαπραγματεύσεις. Μπορώ να, θα μπορούσα να σας πω κι άλλα, αλλά θα ήθελα να σταματήσω εδώ. Εν συντομία για την ανατολική γειτονία, για το θέμα της Ουκρανίας, της Μολδαβίας και της Γεωργίας, ανέκαθεν ε, έλεγα ε, για τις χώρες αυτές και εξακολουθώ να το λέω, έχουμε τις συμφωνίες ε, σύνδεσης της ε, FDA και οι τρεις αυτές ε, χώρες έχουν κυριολεκτικά ξεκινήσει να αξιοποιούν αυτές τις δυνατότητες. Και κατά την άποψή μου, εκεί θα πρέπει να δοθεί η εστίαση αυτές οι δυνατότητες συνολικά να αξιοποιηθούν. Αυτό κατά πρώτον οδηγεί στο να διευκολυνθεί η οικονομική ανάπτυξη. Επίσης βλέπουμε ότι ο όγκος του εμπορίου με τις τρεις αυτές χώρες ε, και την Ευρώπη έχει αυξηθεί σημαντικά. Ειδικότερα από αυτές τις τρεις χώρες, από αυτές τις τρεις χώρες προς την Ευρώπη, ε, οι οποίες ακολουθούν και τα, ευρωπαϊκά, τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά στάνταρ και καλό θα ήταν ε, Καλό είναι που αυτές οι χώρες είχαν, έχουν και είχαν φυσικά αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο, αλλά υπάρχουν δυνατότητες. Οπότε πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτή την κατάσταση, το να σταθεροποιηθεί, να υπάρξουν υποδομές. Πριν λίγα χρόνια εγώ υποστήριξα το ότι πρέπει να καταργηθούν τα τέλη περιαγωγής. Ε, συζητήθηκε και εδώ. Καλό είναι να γίνει αυτή η συζήτηση. Σκεφτείτε, στην Ευρώπη χρειάστηκε 10 χρόνια για να το καταφέρουμε. Ε, κάναμε και ένα πρώτο βήμα στα Βαλκάνια έχουμε και εμπειρίε με το πώς πρέπει να κινηθούμε με αυτό το θέμα, αλλά φυσικά η πρόκληση είναι ότι εδώ έχουμε να κάνουμε ε, με διάφορους που προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν, οπότε πρέπει να βρούμε μια μέση οδό. Ένα από τα deliverables είναι τα τέλη περιαγωγής να καταργηθούν εντός της ε, περιοχής αυτής, αλλά ο απότερος στόχος είναι όπως ε, και για τα Δυτικά Βαλκάνια να τα μειώσουμε μεταξύ ε, των περιοχών αυτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την Λευκορωσία πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερη συζήτηση. Εδώ στόχος θα ήταν να έχουμε κάποιες προτεραιότητες για την εταιρική σχέση, αλλά εδώ σίγουρα δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Πρέπει να δούμε πώς θα καταφέρουμε να βρούμε μια λύση και σε σχέση με το πυρηνικό εργοστάσιο στο Όστροβιτς για τον Νότιο. Ε, ιδιαίτερη προσοχή για την Τινησία. Υποστηρίζουμε τη χώρα αυτή εδώ και μερικά χρόνια με 300 εκατομμύρια ετησίως. Ε, ε, κάθε χρόνο αγωνιζόμαστε ώστε αυτά τα κονδύλια να χρησιμοποιούνται σωστά και αποτελεσματικά. Η τρέχουσα πολιτική κατάσταση δεν συμβάλλει ε, στο να απλουστεύσει αυτή την πρόκληση. Ένα είναι σημαντικό. Αυτή η χώρα πρέπει να υποστηριχθεί έντονα στη δημοκρατική της εξέλιξη και η βοήθεια αυτή ε, ε, πρέπει να αντιγραφεί και για την Αίγυπτο. και εδώ θέλουμε να υποστηρίξουμε ειδικότερα την κοινωνία των πολιτών, το κοινοβούλιο και τις σχετικές εργασίες, η κοινοβουλευτική εργασία να, οι κοινοβουλευτικές εργασίες να ενισχυθούν και στην τομέακη πολιτική να υπάρξει περισσότερη αποτελεσματικότητα. Είναι και δικό μας συμφέρον. Προσπαθούμε δηλαδή να δράμε στοχευμένα με απόλυτη συνείδηση των δυνατοτήτων που έχουμε και των ορίων. Ανέκαθεν έλεγα ότι η Αίγυπτος είναι δίπλα στην ε, Τουρκία και η Ουκρανία είναι η σημαντικότερη γειτονός χώρα της Ευρώπης ε, Οπότε χρειάζεται κάποιος χρόνος για να σας αναλύσω την όλη κατάσταση. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία, ειδικότερα από όσους τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν εδώ ε, και ως πρόεδροι και σε άλλες θέσεις. Πολλοί από εσάς δραστηριοποιηθήκατε ε, στην περιοχή και με βοηθήσατε να σταθεροποιήσουμε κάπως περισσότερο, όπως λέω εγώ συνήθως, τα πράγματα. Και αυτό ήθελα να τονίσω εγώ θα εγκαταλείψω τη θέση μου σε δύο εβδομάδες, ε, όπως ελπίζουμε, ε, αλλά πολύ ειλικρινά ε, θα παραμείνω σε στενές σχέσεις μαζί σας, παρότι θα αναλάβω καινούργια καθήκοντα. Ευχαριστώ. Αγαπητέ Ιωάννης Χάν, Ε, το χειροκρότημα το έδειξε. Είμαστε ευγνώμονε ε, στην Επιτροπή μα για τη δεσμευσή σα ε, μέρα και νύχτα τα τελευταία πέντε χρόνια. Και αυτό που είπατε, το αισθανόμαστε και εμεί για τον Επιτροπό μα, ο οποίο συχνά ερχόταν εδώ και μα μιλούσε στην Επιτροπή μα. Ακούσαμε πολλέ ερωτήσει, κάποιε απαντήσει. Θα μπορούσαμε να έχουμε άλλε τόσε και για τον διάδοχο του Γιωχάνε Χάν. Είναι πολλά τα θέματα όσον αφορά την νοτιοτρική σχέση στα Βαλκάνια που θα πρέπει να συζητηθούν. Ξανά, Ιωάννης Χάν, σας ευχαριστούμε θέρμα. Περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ε, το οποίο θα γίνει και κλεισμένο των θυρών. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω όσους δεν έχουν το δικαίωμα να βρίσκονται εδώ, να εγκαταλείψουν την αίθουσα και γρήγορα παρακαλώ. Ακούω ε, και συζητήσεις φωναχτά. Όσο πιο ήρεμα και γρήγορα τόσο το καλύτερο.